Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie, ale jak Państwo zapewne zauważyli, myśmy cały czas byli na sali. Καλημέρα. Ε, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι είμαστε εδώ. Καλά σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά στην συνεδρίασή μας που θα κρατήσει δύο μέρες, σήμερα και την Πέμπτη. σε δύο μέρη η συνεδρίαση. Πλήρω το πρόγραμμά μας. Και μια και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις επειδή είναι Δευτέρα, να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, καλωσορίζοντας μια συνάδελφο που ήρθε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και που αυτό το καιρό έχει αναλάβει σημαντικά πολιτικά καθήκοντα και σημαντικό πολιτικό αξίωμα στην πατρίδα της. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Και επειδή σήμερα το απόγευμα απουσιάζει ο κύριος Μισελ Νταντάν, ο συντάκτης γνωμοδότης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα την πολιτική συνοχή στις ορεινές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνω η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σημείο αυτό να αναβληθεί για την Πέμπτη το πρωί. Επίσης θα προσπαθήσουμε το σημείο 7 να το εξετάσουμε το 13, άμα το επιτρέψει ο χρόνος. Αυτά για την Πέμπτη. Επίσης, λόγω απουσίας ε, τη εισηγήτρια ε, στι συνεχείς διοργανικέ διαπραγματεύσει για τα μέτρα προστασία της υγεία των φυτών τη, κυρία Μακιντάερ θα πρότεινα την δική της παρουσίαση για την κατάσταση και τις εξελίξεις στο θέμα αυτό ε, να την αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Και με αυτές τις δύο αλλαγές και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα έλεγα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας να μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου η συνεδρίαση και επίση υπάρχει διερμηνία από και προς 18 γλώσσες με εξαίρεση στα δανέζικα, αισθανικά, μαλτέζικα, σλοβακικά, κροατικά και κελτικά. Έχετε λάβει προς έγκριση τα πρακτικά της 1 ης Οκτωβρίου του 2015. Μέχρι το πέρας συνεδρίες δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα. Και περνάμε στο τέταρτο σημείο της ημερήσης διάταξης που είναι και το πρώτο ουσιαστικό σημείο, πολύ σημαντικό της ημερήσης διάταξης και αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για τη διανομή οποροκυπευτικών, μπανάνων και γάλακτος στα σχολεία. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Μάρκ Ταραμπέλα. Η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Γεωργίας είναι η αρμόδια κατ' Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ταραμπέλα θα μας παρουσιάσει τις εξελίξεις της 20 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη, ο πρώτος τριμερής διάλογος για το πρόγραμμα αυτό διανομής απορροκριστικών στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αυτό θα ήθελα να τονίσω γιατί αφορά τη δωρεάν διανομή υγιεινών γεωργικών προϊόντων στα σχολεία για τα παιδιά με κοινοτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα ε, εν μέσω κρίση. Και έχει και παιδαγωγική αξία αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει όμω ένα πρόβλημα με το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, γιατί το Συμβούλιο δεν δέχεται τη συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, με βάση το άρθρο 43 πάραγραφό 2 και προτιμά να μονοπολίσει την αρμοδιότητα για το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Αυτά όμω πιο διεξοδικά θα μας, θα τα, μας τα αναλύσει ο εισηγητής μας, ο κύριος Ταραμπέλα, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τις άκρες προσπάθειες που καταβάλει στο θέμα αυτό. Έχει πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό η ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του βουλευτών στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις του Συμβουλίου, του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και των σχεδόν εισηγητών και των συντονιστών. Μάλιστα, στείλαμε σχετική επιστολή για το θέμα αυτό στον πρόεδρο Σούλτς, σε συμφωνία με τον εισηγητή και τους συντονιστές, ζητώντας από τον πρόεδρο Σούλτς να διαβιβάσει τις ανησυχίες μας ε, στα υψηλότερα κλεμάκια του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής. Και θα ακούσουμε τώρα τον εισηγητή μας τον κύριο Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή σας επιμείνατε και εσείς το γεγονός ε, ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό για τα παιδιά, για τα σχολεία, για τη δημόσια υγεία και ακριβώς λόγω της σημασίας του, όπως είπατε και εσείς, έγινε ένας πρώτος τριμερής διάλογος ε, στις 20 Οκτωβρίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα και θα πρέπει εδώ ίσως λίγο να παρακάμψουμε και το πρωτόκολλο και τα έθιμα και τους ε, κανόνες. Ε, θα ήθελα ο καθής από τους και εισηγητές και από τις πολιτικές ομάδες που ήταν ε, παρόντες να εκφράζουν με μία φωνή την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι η νομική βάση επί της οποίας θέλει να εργαστεί το Συμβούλιο είναι μη αποδεκτή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 43.3 προβλέπει ότι το Συμβούλιο έχει όλα τα δικαιώματα στα θέματα αυτά και την ευελιξία στα προγράμματα και τον προπολογισμό και τον κατάλογο των προϊόντων. Ε, υπάρχουν βέβαια και κάποια προϊόντα στα οποία υποχωρήσαμε. Είναι απαράδεκτο λοιπόν αυτό. Είμαστε ενωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες που υπέγραψαν την επιστολή που αποστέλουμε στον πρόεδρο Μαρτίν Σούλτς για να ε, ε, ασχοληθεί με το θέμα αυτό για την άποψη αυτή του Συμβουλίου ότι το άρθρο 43.3 ε, από, εφαρμόζεται γενικώ. Υπάρχει ακόμα υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία λέει ότι το άρθρο 43.3 δεν προβλέπει ούτε συναπόφαση ούτε και κάποιο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση σε κάποια ζητήματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα τα πάντα να καλύπτονται από το άρθρο 43.2 που μας επιτρέπει να έχουμε συνεπόφαση. Υπάρχουν όμως τρία βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συναπόφαση. Τα κριτήρια διανομής των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να αποτελεί συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας πω ότι υπάρχει μια συνολική συμφωνία που ε, επιτρέπει να χρησιμοποιούνται ιστορικά κριτήρια και κάποια αντικειμενικά κριτήρια και να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα επιλέξουν και στο Συμβούλιο. Επίσης, η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των προγραμμάτων είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να μπορούμε να έχουμε γιατί στο Συμβούλιο ξέρετε τι γίνεται για να συμφωνήσουν ε, επειδή υπάρχουν εθνικά συμφέροντα, τα οποία ίσως εκφράζονται πολύ περισσότερο στο Συμβούλιο από ό,τι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να υπάρχουν κάποια ε, προγράμματα τα οποία να μην έχουν καθόλου κονδύλια προς όφελος κάποιων άλλων προγραμμάτων. Για παράδειγμα, στην Φιλανδία καταναλώνεται πολύ γάλα, αλλά ελάχιστα φρούτα. Ε, χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Φιλανδίας, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά σίγουρα είναι προς το συμφέρον τους να υπάρχει και πρόγραμμα για τα προκυπευτικά και για τα φρούτα. Και να μην πούμε ότι δεν θα έχουμε φρούτα για να ενισχύσουμε το γάλα στη Φιλανδία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και εμεί ε, αρμοδιότητα εδώ. Και τέλο υπάρχει και το θέμα του προπολογισμού. Ε, τον προπολογισμό μπορεί να τον αποφασίσουμε φέτο και αν το Συμβούλιο πει ότι του χρόνου θα κάνουμε οικονομίε στο θέμα αυτό και θα βάλουμε τον προπολογισμό στο 10% ή στο 0%, ε, θα πρέπει να έχουμε και εμεί λόγο. Πρέπει λοιπόν να συναποφασίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό δεν επέδειξα καμία ευελιξία, δεν ξεκίνησε διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο του θέματο, εάν το Συμβούλιο δεν επανέλθει με ε, νέα θέση και τουλάχιστον τουλάχιστον αυτά τα τρία ζητήματα να ε, καλύπτονται με βάση το 43-2, δηλαδή με βάση συναπόφαση. Συγγνώμη, χτυπάει το τηλέφωνο γιατί πρέπει στις 3 ε, και 4 να μιλήσω για τις ε, ε, δημόσιες συμβάσεις στην ΙΜΚΟ. Αυτό όμως το θέμα με ενδιαφέρει περισσότερο κύριο πρόβλημα, Πρόεδρε, και θα φύγω μόλις ολοκληρωθεί αυτό. Ζητώ λοιπόν, στις 11 Νοεμβρίου είναι και η κυρία Μίλλερ εδώ που είναι σκιώδη συζήτητρια από πλευράς φιλελευθέρων αλλά ελπίζω να συμφωνούν. Θα κάνουμε μια συμφωνία στις 11 το πρωί γιατί θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου ο δεύτερος τριμερής διάλογος το απόγευμα στις 2 η ώρα στο Συμβούλιο και ελπίζω το, το Κοινοβούλιο να τηρήσει την ίδια στάση διότι Υπάρχει και εσωτερική εμπειρία που γνωρίζουμε από το Κοινοβούλιο. Σε κάποια άλλα θέματα δεν, δεν ξέρω αν θυμάστε. Τελικώ είπαμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και θα δούμε τη νομική βάση αργότερα και μετά στο τέλος καταλήξαμε σε συμφωνία και μας είπαν ότι ή αυτή τη νομική βάση ή τα εγκαταλείπουμε όλα. Εγώ δεν θέλω να το παίξω αυτό το παιχνιδάκι, επομένως ε, ε, Ξέρω ότι θα συναντήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συναντήσουμε και το Συμβούλιο πριν, ε, αλλά προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρήσει αυστηρή στάση και να πει ότι δεν διαπραγματευόμαστε εάν δεν έχουμε ως νομική βάση το άρθρο 43.2. Να είναι λοιπόν συναπόφαση για τον προπολογισμό, για τα κριτήρια διανομή και για τη μεταφορά κονδυλίων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Αυτά λοιπόν τα τρία θέματα που μα αποσχολούν και από εκεί και πέρα απευθύνομαι σε εσά. Θα ξανάρθω εδώ να σα πω τα αποτελέσματα του τριμερίου διαλόγου, αλλά ελπίζω να έχουμε ομόφωνη θέση ε, ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι ο μόνο τρόπο να έχουμε μια έκθεση η οποία θα είναι ισορροπημένη και επίσης να υπενθυμίσω ότι εδώ δημιουργείται προηγούμενο. Εάν δεχτούμε τώρα το 43-3 για κάθε θέμα θα θέλουν να εφαρμόσετε το 43-3 Και υπενθυμίζω ότι για θέματα προπολογισμού θα πρέπει τουλάχιστον το Κοινοβούλιο να δίνει την άποψή του και να γίνει σεβαστό αυτό. Δεν δώσαμε μάχη για να έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνα που να μας δίνει στην απόφαση, στη Γεωργία τουλάχιστον, που γνωρίζουμε τι συνέβαινε στο παρελθόν, για να μας την ε, ε, εμφανίζουν σε κάθε θέμα ε, θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα πριν από τα Χριστούγεννα στη διάρκεια της Λουξεμβουριανής Προεδρίας αλλά όχι με κάθε τίμημα και ελπίζω ε, να γίνει δεχτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπενθυμίζω ότι έκανε πολύ καλή πρόταση στην αρχή και εμείς απλώ κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και έχω περισσότερες αμφιβολίες για την πρόταση του Συμβολίου. Ελπίζω λοιπόν αυτή η θέση να γίνει δεκτή και να την υποστηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Περιμένω και τα σχόλιά σας έτσι. Πρέπει να φύγω για τη ΜΜΚΟ αλλά δεν θα φύγω έτσι. Έχουμε συζήτηση εδώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βουλευτά. Όπως είπατε κι εσείς, θέλετε να ακούσετε τις απόψεις των συναδέλφων. Δώσω το λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Μάρκ Ταραμπέλα για το έργο του, γιατί ήταν εξαιρετική η προσπάθειά του και διαμόρφωσε ένα πολύ καλό περιεχόμενο στην έκθεσή του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή και στα θέματα της υγείας. Και επίσης ε, χαιρετίζουμε το διάβημά του ε, και τη θέση που κράτησε κατά την έναρξη του τριμερούς διαλόγου. Γιατί όπως δεν θα πρέπει πάση θυσία να κάνουμε ε, υποχωρήσει, αλλά πάση θυσία να αποφύγουμε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο εδώ. Η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και θα δεν αφήσουμε να μα τριμώχνουν αριστερά και δεξιά. Από τη μια να ροκανίζει τη βασική πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέροντα πολλά σημεία στι κατεξιοδότηση πράξη και από την άλλη να ροκανίζει τι αρμοδιότητέ μα στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να εμείνουμε στεναρά και να διατρανώσουμε τις εξουσίες μας και τις αρμοδιότητές μας επιδεικνύοντας αλληλεγγύη. Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου προς τον εισηγητή στον αγώνα που δίνει και δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε με τίποτα και να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την άποψή μας υπέρ των συμφερών των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, για τα τρία σημεία, το θέμα του προϋπολογισμού, του κριτηρίου κατανομής και της μεταφοράς μεταξύ των προγραμμάτων, αυτά τα τρία σημεία είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να μείνουμε αμήλικτοι και αδιάλακτοι, γιατί από τη θέση μας σε αυτά τα τρία θέματα θα εξαρτηθεί το μέλλον των διαπραγματεύσεων στο διμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Μάρκ Ταραμπέλα για τη στάση που έχει κρατήσει ως τώρα η Περιμόνα. Φυσικά τον υποστηρίζουμε, είμαστε στο πλευρό του και επιμένουμε στις βάσεις επί τις οποίες εργάστηκε. Εδώ βλέπουμε ότι κουράστηκε πολύ για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μια καλή θέση, ειδικότερα στο θέμα της υγείας και της εκπαίδευσης ε, που θα προσφέρουμε στα παιδιά μας. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι σωστή και εμείς ε, θα συμμετέχουμε από κοινού και θα λάβουμε μέρος και στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ για την δουλειά σας λοιπόν. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μάρκ Ταραμπέλα για τη θέση που έχει λάβει. Έχει ε, μια θέση πολιτική με την οποία συμφωνώ πλήρως ε, σε διάφορα σημεία. Η ε, γερμανική η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μια κάπως διαφορετική θέση. Παρ' όλα αυτά εγώ παρόλο που είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Γερμανίας έχω και μια ευρωπαϊκή ευθύνη και λόγω αυτής της ευρωπαϊκής ε, ευθύνης τον υποστηρίζω πλήρως. Να πω τέλος ότι ε, θα πρέπει να βγάλουμε έναν κανονισμό ο οποίος ε, δεν θα είναι καθόλου γραφειοκρατικός. Θα πρέπει εδώ ε, να έχουμε υπόψη μας ότι τα χρήματα που δίνονται δεν είναι τεράστιο ποσό, είναι λίγα χρήματα και γι' αυτό θα προσπαθήσω να συζητήσω και με τις ομάδες, ε, τις πολιτικές, ώστε να έχουμε μία κοινή θέση στο Κοινοβούλιο, να έχουμε έναν, ε, μία ενωμένη θέση απέναντι στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Δεν ακούσαμε το όνομα του επόμενου μιλητή δυστυχώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Ταραμπέλα και να τον συγχαρώ θερμά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες γιατί είναι πολύ σωστή έκθεση, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Βέβαια, φοβούμε ότι χάνουμε μια λαμπρή ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία και αυτό με απογοητεύει. Γιατί δεν διευρύνουμε τα προγράμματα διανομής ε, ε, στα σχολεία σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το μέλι ή οι ελιές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να παρουσιάσει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σχετική πρόταση. Έχουμε ένα χρόνο περίπου καθυστέρηση δυστυχώς είχαμε πει να ε, παρατείνουμε το πεδίο εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων για τα σχολεία και να περιλάβουμε και άλλα προϊόντα, όπως σας είπα, το ελαιόλαδο, τις ελιές και το μέλι. Δυστυχώς, ε, να είχαμε ζητήσει να συνταχθεί σχετική έκθεση για την επέκταση του προγράμματος, ποτέ δεν έγινε. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα και είναι κρίμα που τα, τα προϊόντα που ανέφερα αποκλείστηκαν από τα προγράμματα διανομής. Και μιλούμε για υγιεινά προϊόντα, πολύ ωφέλιμα για την υγεία των παιδιών, που το, ούτως ή άλλως αποτελούν στοιχείο το, της παραδοσιακής διατροφής, κυρίως των νότιων χωρών της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να ξανατονίσουμε την ανάγκη να συμπεριλάβουμε και τα προϊόντα αυτά που σας ανέφερα στα προγράμματα διανομής υγιεινών γεωργικών προϊόντων στα σχολεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δερνανό. Oui, ναι κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ε, το είπα μάλιστα, δεν χρειάζεται να επανέλθω. Θα συμφωνώ και εγώ να σε χαρώ τον κύριο Ταραμπέλα για ό,τι έκανε. Στο θέμα της οργάνωσης του προγράμματος, ε, τα προγράμματα είναι εξελίξη αλλά το θέμα του προπολογισμού είναι κάτι ε, επί του οποίου πρέπει να έχουμε και εμείς άποψη. Στις 5 ε, η ώρα θα ξεκινήσει η συνδιαλλαγή και θα πρέπει να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτό το πρόγραμμα για τα φρούτα και τα απορροκυπευτικά και στον προπολογισμό και εγώ ως συντάκτης της είχα ζητήσει να υπάρχει ένα ποσό το οποίο να μην είναι αμεληταίο για αυτά τα φρούτα και τα απορροκυπευτικά και ταυτόχρονα ο Μάρκ Ταραμπέλα ε, πιέζει για το θέμα των προγραμμάτων, επομένως θα πρέπει και το θέμα του προπολογισμού να ε, το λάβει αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράν. Oui, Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σύμφωνο και εγώ με τις απόψεις και η ομάδα μας, η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, ε, υποστηρίζουμε την ε, πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, Γεωργίας του Μαρκ Ταραμπέλα, εξ ονόματος των βουλευτών, που θέλει να προασπίσει τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου σε αυτά τα προγράμματα ενίσχυσης. Πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά μόνο του χωρίς την ε, ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και σήμερα δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη, να μην μάλλον λάβουμε υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Υπερψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση του Μαρκ Μπέλα για τρεις λόγους, για την καταπολέμηση της κακής διατροφής, ε, υπέρ της υγείας και της βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Äh, Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την υποστήριξη της ομάδας μου για την πρόταση του ε, Μάρκ Ταραμπέλ. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι περιλαμβάνει όλα τα σημεία που μας ενδιαφέρει. Άκουσα από τα, ε, διάβασα από τα ε, πρακτικά ότι το Συμβουλίο δεν είναι ολόκληρο. Είναι κάποια κράτη-μέλη που στην ουσία συμμετέχουν Και επειδή είναι και κάποιος δικός μας ε, ε, σύμμαχος εκεί, ε, την ίδια πολιτική ομάδα, καλό θα είναι να τους πούμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι και πρέπει και στην πατρίδα μας αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Όταν μιλάμε για εκπαιδευτικά ιδρύματα και για διατροφή, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε προγράμματα τα οποία δεν θα θέτουν τίποτα άλλο παρά μόνο την εκπαίδευση και την διατροφή ε, στο προσκήνιο. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον για κάποιον που είναι λίγο καιρό εδώ και παρατηρεί τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται ή που απαιτείται να παίζονται για να ακουστεί το κοινοβούλιο. Για το θέμα αυτό καθεαυτό, το βλέπω κάπως περίεργο που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο στην ουσία οργανώνει τι θα φάνε τα παιδιά στο πρωινό τους όταν υπάρχουν εξαιρετικά τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα μπορούσαν αυτά να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό στην ουσία που γίνεται είναι προπαγάνδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Χρειάζεται μεν η θετική προπαγάνδα, το λέμε αυτό, γιατί ενώ λέμε ότι ταΐζουμε τα παιδιά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατάμε υγιή, ε, στο κρατικό επίπεδο τα παιδιά ε, προσπαθούν να πάρουν πρωινό μέσω των, μέσω των γονιών τους. Ε, στην ουσία αυτό που γίνεται όμως είναι ε, να κοινωνικοποιούνται τα χρέη των τραπεζών μέσα από αυτό στην ουσία γίνεται μια κλοπή στους ανθρώπους και μέσα από αυτό ε, και, μέσα, και σε αυτό το τομέα περνάει αυτό. Εξαιρετικά παιχνίδια πραγματικά τα απολαμβάνω. Πριν ολοκληρώσουμε τον γύρο των ομιλητών, θα δώσω το λόγο στην κυρία Σένερα και τέλος στον εισηγητή μας και πάλι στον κύριο Ταραμπέλα. Κυρία Σένερα. Με το πρόγραμμα αυτό θεωρώ ότι ασχοληθήκαμε εκτενώς εδώ. Κάναμε μεγάλες προσπάθειες και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοια προγράμματα ε, στήριξης ε, για να προωθήσουμε την αξία της διατροφής ε, και να εξοικειώσουμε τα παιδιά με το από πού προέρχονται τα τρόφιμα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μας κοροϊδεύει το Συμβούλιο. Και γι' αυτό θα ήθελα να εκδηλώσω την αμέριστη υποστήριξή μου στις προτάσεις του συγγετού μας του κυρίου Ταραμπέλα. Θα ξαναδώσω το λόγο στον συντάκτη μας, τον κύριο Ταραμπέλα, γιατί στον εισηγητή μας, τον κύριο Ταραμπέλα, γιατί πρέπει να πάει και σε άλλη συνεδρίαση και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιώστε. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την ομόφωνη υποστήριξη στην στάση που θέλω να τηρήσω, διότι δεν το είπα, μεν, αλλά στον προηγούμενο τριμερή διάλογο η πρόταση που έγινε και από πλευρά Συμβουλίου και λίγο και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε ως προς το περιεχόμενο και να δούμε την νομική βάση αργότερα. Εγώ ε, προτείνω να τηρήσουμε αυτή την αυστηρή στάση και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ε, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον και ε, χάνει την εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να γίνεται σεβαστό και δεν θα πρέπει να μας ε, στερούν αρμοδιότητε. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε προηγουμένως στον κατάλογο των προϊόντων. Υπάρχει ένα συμβιβασμό εδώ, αυτό είναι σαφέ και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ούτε το Συμβούλιο θα έχει δίκιο εναντίον του Κοινοβουλίου, ούτε το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι έχει και ένα συμβιβασμό, δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι με βάση ακριβώς ε, τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουμε κάποια προϊόντα, θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε, δεν έχουμε πει τίποτα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, δεν μπορούμε να τα ξανανοίξουμε όλα γιατί υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι λιγότερο υγιεινά από όποια υπόλοιπα. Σίγουρα λοιπόν θα ξαναγίνει συζήτηση για τα θέματα αυτά. Θα συζητούμε με τους κοιόδες συζητητέ. Ούτως ή άλλως θέλω να συζητούμε εκ προημίου για να υπάρχει μια στεναρή στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε τουλάχιστον στο συμβιβασμό στον οποίο θα καταλήξουμε στο τέλος να υπάρχει και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Φλάναγκα, ε, τι να σας πω κύριε Φλάναγκα, κατάγεστε από την Ιρλανδία, όπου το ποσοστό της παχυσαρτυχίας των παιδιών είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύντομα το 80% των μικρών Ιρλανδών δεν θα μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο ή ράγμπι γιατί είναι παχύσαρκα. Αν λοιπόν αφήσουμε στα κράτη-μέλη την ελευθερία να ρυθμίσουν όλα τα προβλήματα, τότε η Ευρώπη ε, θα πρέπει και αυτή να προσπαθεί με έναν τρόπο να συνεισφέρει και αυτή το λιθαρότητα της. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά έχει και η Ευρώπη αρμοδιότητα για να λύσει το πρόβλημα τη δημόσια υγεία. Και σα το επαναλαμβάνω, στην Ιρλανδία το πρόβλημα τη παιδική που έχει παχυσαρκίας είναι από τα πιο σοβαρά. Πώ μπορούμε λοιπόν να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μα ε, να διατρέφονται σωστά. Και υπάρχουν 24-28 χώρες που κατανοούν πολύ λιγότερα οπορακυπευτικά και φρούτα με βάση τις συστάσεις του ΠΟΗ. Και η Ιρλανδία έχει τις χειρότερες επιδόσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστούμε κύριε Φλάνναγκαν, λοιπόν που θα μας αφήσετε λίγο και το ελεύθερο στο θέμα αυτό. Εμείς. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε στο πλευρό σας ε, κύριε Ταραμπέλα. Φάνηκε αυτό από τη στριπτική πλειοψηφία των ομιλητών που τάχθηκε υπέρ α, ε, ε, του εισηγητού και μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να κερδίσουμε. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν βρίσκεται στην αίθουσα, αλλά δεν βλέπω κανέναν. Όπως ξέρετε, στείλαμε επιστολή με υπογραφή του υποφανεμόνου Προέδρου, του κ. Ταραμπέλα, των συντονιστών. Αποστήλαμε επιστολή λοιπόν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Σούλτς, για να διαβιβάσει την άποψή μας στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Γιούνκερ. Έχει αντίγραφα η γραμματεία, αν θέλετε, να ενημερωθείτε σχετικά. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το σημείο 5, όπως είπα, το αναβάλαμε για επόμενη συνεδρίαση. Α, ο κύριος Φλάνακαν, συγγνώμη. Αλλά παρακαλώ όχι αντιπαραθέσεις τώρα, όχι διεξυπισμούς. Δεν θα μπω σε μεγάλη συζήτηση. Είχαμε πολύ καιρό προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσαν για μας τόσο καλά. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Υπάρχουν προβλήματα παχυσαρκίας στην Ευρώπη, δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να, να είναι κάποιος δακτυλοδεικτούμενος. Δεν είναι δίκιο, γιατί τελικά ο καθένας είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι είναι η Ευρώπη ή η Ιρλανδία ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Αυτό που ε, ευθύνεται είναι η Coca-Cola, οι μαζικές πολυεθνικές ε, που συμβαινει αυτο αυτο που ευθυνεται ειναι η κοκακολα οι χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτό το σώμα και η δική τους ατζέντα το να ε, ρίχνουν αυτά τα πράγματα με το ζόρι στο στόμα μας στην ουσία μας κάνει παχύσαρκους και αν δεν μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτούς δεν θα το κάνουμε μέσω από το TTIP φυσικά ε, ε, αν θέλετε κάτι να κάνετε λοιπόν κάντε το εκεί μην πάτε όμως ως ιεροκήρυκες να κάνετε κήρυγμα σε ανθρώπους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να τους λέτε τι πρέπει να φάνε για το πρωινό τους. Εμείς σίγουρα πρέπει να τα πάμε καλύτερα στην Ιρλανδία. Εγώ η ίδιος ε, κάνω μαραθώνιο και εξασκούμε και δίνω το παράδειγμα. Ελπίζω και εσείς να κάνετε το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να βελτιώσουμε το πρόγραμμα. Και αυτά που μόλις είπε ο κύριος Φλάναγκαν αποδεικνύουν ότι πρέπει να βελτιωθεί το πρόγραμμα και νομίζω ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προς τη σωστή άγουσα. Θα τα καταφέρουμε με την υποστήριξη του κ. Φλάναγκαν και χωρίς την υποστήριξή του. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Σας ευχαριστούμε. Ε, νομίζω ότι μετά τα τελευταία σχόλια φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη σύγκληση των απόψεων. και έχει ο κύριος Φλάναγκαν. Μακάρι να είχα και εγώ το σώμα ε, του κυρίου Φλάναγκαν, γιατί πραγματικά είναι σε μεγάλη φόρμα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο. Okay. Okay. Εκτός μικροφόρου, δυστυχώς το σχόλιο του κ. Φλάναγκαν. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 6, με θέμα τη βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Γιάνν Χαϊτεμα. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας ε, από την ομάδα των φιλελευθέρων ήταν δική της η πρωτοβουλία και ο κύριος Χάιτεμα θα εκπονήσει την έκθεση αυτή ίδιας πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η καινοτομία και η ανάγκη της βελτίωσής της ε, για την οικονομική ανάπτυξη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει ολόκληρο τον κλάδο της ευρωπαϊκής γεωργίας. Πολλές συζητήσεις γίνονται για την καινοτομία στη Γεωργία. Για πολλά χρόνια ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, τις καινοτόμες γεωργικές πρακτικές που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και μάλιστα η, η πατρίδα του κ. Χώτημα είναι πρωτοπόρο σε τέτοιες καινοτόμες γεωργικές πρακτικές και μάλιστα από το χρόνο τον Ιανουάριο θα αναλάβετε και την Προεδρία Οπότε ελπίζω να προωθεί ακόμη περισσότερο το θέμα στη διάρκεια τη Ολλανδικής Προεδρίας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή μα τον κύριο Χέιτεμα, για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως ε, ε, και εγώ όπως και εσείς φαντάζομαι θεωρούμε πως ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας είναι εξαιρετικός, ε, είναι προοδευτικός και το πιο σημαντικό είναι ε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κερδίσουμε από αυτόν τον τομέα και είναι πιο απίστευτο ακόμα. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Χρειαζόμαστε σύμφωνα με το ΦΑΒ 70% αύξηση στην παραγωγή τροφίμων για να ταΐσουμε πάνω από 9 εκατομμύρια ε, άτομα ακόμα και στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουμε αύξηση 23% στα σιτηρά. Εξαιτίας ε, και των αλλαγών στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ε, λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξης και του πλούτου στον κόσμο, υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση στις πρωτεΐνες όπως το τυρί, το γάλα και τα λοιπά και το κρέας. Έτσι λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον μας και να αντιμετωπίσουμε και την αλλαγή του κλίματος που οδηγεί και σε αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Έτσι λοιπόν η μεγάλη καταστροφή μπορεί να διαφαίνεται, αλλά η λύση είναι απλή. Πρέπει να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα και με έξυπνο τρόπο. Η μόνη καλή λύση λοιπόν είναι η ενίσχυση της καινοτομία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, από τότε που ξεκίνησαν οι άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη, πάντοτε έψαχναν για καλύτερες λύσεις στην παραγωγή. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το σταυροδρόμι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε για το μέλλον μας. Θα πάμε προς, τα μπρος ή προς τα πίσω, προς το παρελθόν. Η καινοτομία ε, είναι ε, κάτι που χρειαζόμαστε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση ενώπιό μας ε, και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι σωστό για τη διοργία του, του μέλλοντος αυτός ο κατάλογος ε, που θα έπρεπε, των καινοτομιών που θα έπρεπε να γίνουν είναι τεράστιος. Ε, οι νέες ε, λύσεις της τεχνολογίας και των δεδομένων οδηγούν σε μηχανήματα που μπορούν να καλλιεργήσουν στην, τη γη ακόμα και με ακρίβεια δύο εκατοστών. Μπορούμε έτσι να μειώσουμε την ανάγκη για λίπασμα, για κατανάλωση νερού, και για μεγάλες εκτάσεις. Ε, υπάρχει νέος ε, τρόπος ανάπτυξης πρωτεϊνών, όπως για παράδειγμα μέσω εντόμων, ε, και υπάρχει και άλλος τρόπος αξιοποίησης της κοπριάς έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα λιπάσματα. Δεν χρειάζεται να καίμε ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή των Όμω Όμως η κοινή γεωργική πολιτική δεν επικεντρώνεται αρκετά στις νέες αυτές εξελίξεις που θα έπρεπε να είναι ψηλά στην Ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη ενώ τώρα οι επιχειρηματίες στη γεωργία αντιμετωπίζουν παροχημένους και δύσκολους κανόνες. Βέβαια οι αναλλαγές γίνονται βήμα-βήμα. Αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα ως έρχεται. Γι' αυτό χρειάζομαι και την βοήθειά σας συνάδελφοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για πληροφορίες ε, στο γραφείο μου. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, δυστυχώς όμως κάποιοι από εσά δεν έχετε ακούσει τίποτα. Έτσι λοιπόν συμμεριζόμαστε τα προβλήματά σας ε, και θέλουμε μερικά από αυτά, ό,τι αφορά στη χώρα σας, να το εντάξουμε στην προσπάθειά μας. Τι είδους νομοθεσία θεωρείτε ότι είναι προβληματική, πού βλέπετε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή γεωργία. Πραγματικά αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι επίκαιρη και ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τις καινοτομίε που λαμβάνουν χώρα στη χώρα σας και ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ο κύριος Άλμπερντ Έσταρ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ ε, τον ε, εισηγητή για αυτή την έκθεση. Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα γιατί οι καινοτομίες που θα μας φέρουν πιο κοντά στο μέλλον είναι ε, πραγματικά δυνατόν να συμβούν. Δυστυχώς στην μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη μας τις ε, νέες, μοντέρνες ε, ε, πρακτικές. Υπήρξε λίγη υποστήριξη δυστυχώς. Με κάποιους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, εκπλαγήκαμε πραγματικά όταν συναντηθήκαμε γιατί μας έδειξαν πολύ μοντέρνες τεχνικές. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα ρομπότ το οποίο πηγαίνει μέσα στο ε, χωράφι και βρίσκει εκεί που είναι οι πατάτες ακριβώς που βρίσκονται τα παράσιτα. Μπορεί λοιπόν με 100% ε, να αποφευχθεί ο ψεκασμός αυτών των επιφανειών. Τέτοιες είναι οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Πραγματικά πάντοτε με ε, εντυπωσιάζει πόσο μεγαλώνουν τα τρακτόρ, τα, τα τρακτέρ στη χώρα μου. Ε, ε, συνεχώς ε, ξεκινήσαμε με τα 100, με τα 150, φτάσαμε στα 300 πια. Ε, έχουμε όμως ένα νέο μοντέλο στη χώρα μας με τριαξονικό 50 ύπους, το οποίο μπορεί ανεξάρτητα 24 ώρες το τετράωρο να εργάζεται και να, ε, να βοηθά στην καλλιέργεια της γης. Είναι λοιπόν μια τεράστια ε, ευκαιρία που έχουμε για το μέλλον. Οι τεχνικές μπορούν να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν είναι να βγάλουμε από την καλλιέργεια κάποιες εκτάσεις και να φάζουμε εκεί λουλούδια. Το θέμα είναι να έχουμε πιο σύγχρονες τακτικές και τεχνολογίες για να βελτιώνουμε την καλλιέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε ήμουν φίλος της τεχνολογίας ε, και ακριβώς αυτή η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να είμαστε και φιλικοί προς το περιβάλλον που ακόμα περισσότερο με ενθουσιάζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Εγώ περίμενα λίγα περισσότερα ε, το θέμα της καινοτομίας. Ε, δεν με ε, εξέπληξε αυτό. Κάτι για τα γενετικά τροποποιημένα περίμενα, αλλά δεν είπατε τίποτα. Αυτά που είπατε είναι πολύ τεχνολογικά. Και ε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η εντατική γεωργία ε, δεν ε, ακολουθεί ακριβώς αυτή την κατεύθυνση που θα έπρεπε και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η τεχνολογία, το αναφέρατε πριν, ε, όπως, όσον αφορά το όργωμα. έτσι λοιπόν να πω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, πρέπει πάντοτε να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορούμε και στη γεωργία να έχουμε βιώσιμη ανάκτηση ανάπτυξη και να μεγιστοποιούμε και την παραγωγή. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες ζωικές ε, πρωτεΐνες. Ε, ε, δεν καταλαβαίνω τελικά πώς φτάνουμε σε αυτή την κρίση με το γάλα και γενικά υπάρχουν τόσα πολλά προϊόντα που παράγονται και δεν, και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που θέλουν το Ολλανδικό και το Γερμανικό κρέας ε, και περιμένουν το γάλα της Ευρώπης. Υπάρχει 1,3 ε, ε, δις άνθρωποι που έχουν βασικές ανάγκες και δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει ακριβώς να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της σπατάλης. Χρειάζεται λοιπόν ε, να ασχοληθούμε με την αλυσίδα της οικονομίας, όχι μόνο με την υποδομή, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν ε, τελικά ε, όλο και περισσότερο παράγουμε, αλλά όλο και λιγότερα χρήματα παίρνουν οι γεωργοί που παράγουν. Όλο και περισσότερα κερδίζουν. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι και αυτά μέσα στη μελλοντική μας στάση, μαζί με την καινοτομία και μαζί και με την βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία. Η, τεχνολογία από μόνη της είναι ε, λίγη θα έλεγα. Τα βιώσιμα συστήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το input, το τι μπαίνει, αλλά και με το τι βγαίνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα η βιοπικιλότητα χάνεται με την αντιρρητικοποίηση της γεωργίας. Συμβάλλουμε και σε αυτό. Χωρίς τη βιοπικιλότητα δεν μπορούμε ούτε σωστή γεωργία να έχουμε. Συζητήσαμε επίσης ε, για το τι κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε τη βιοποικιλότητα στην γεωργία έτσι ώστε να έχουμε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις έτσι ώστε ε, να έχουμε μεθόδους που όλο λιγότερα θα θέλουν ως εισρωή και όλα περισσότερα θα βγαίνουν ως εκροή και θα φέρνουν και περισσότερο κέρδος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την εισαγωγή που μας έκανε στην έκθεσή του, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντική για τη συνέχιση της συζήτησης ε, και τους προσανατολισμούς που θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Κάτι όμως που θα πρέπει να μας ε, προβληματίσει πρώτα απ' όλα, όπως φάνηκε και από αυτά που είπαμε, είναι ναι καινοτομία, αλλά στην υπηρεσία ποιας γεωργίας. Ε, εκεί μερικές φορές υπάρχουν διαφορές. Γιατί ο κύριος Χαϊτεμά είπε σωστά ότι αν θέλουμε, θέλουμε να παράγουμε περισσότερο αλλά λιγότερα. Εγώ θα έλεγα να παράγουμε καλύτερα με λιγότερα. Γιατί όταν κάνουμε τον απολογισμό της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, από την ε, έναρξη εφαρμογής της, εγώ θα έλεγα ότι είναι επιτέλους ε, η ώρα να διαρωτηθούμε τι προκάλεσε και ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής, ε, της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και αν όντω εξασφαλίσαμε την επιστημιστική ασφάλεια, αν ε, ε, επιτύχαμε την ποιότητα των τροφίμων, αν εξυπηρετήσαμε τους σκοπούς της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, υπάρχει το θέμα της απερίμωσης ή της φτώχησης των εδαφών, της το θέμα της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ε, το θέμα του ύδατος, ε, το θέμα της απασχόλησης στις τοπικές οικονομίες. Ο Άλπερτες είπε ότι σαγηνέθηκε από τα τρακτέδα που κινούνται από μόνα τους χωρίς οδηγό. Έτσι όμως χάνουμε θέσεις απασχόλησης. Αν είναι αυτόματο το τρακτέρ, δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι η υπερβολική η εφαρμογή των, ε, η εισαγωγή των ρομπότ στη Γεωργία θα μας στερήσει από ανθρώπινο δυναμικό και από εργατικά χέρια. Πήγαμε πέρυσι σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή και βλέπουμε ποια είναι η σχέση της γεωργίας και της απασχόλησης τόπου. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία. Τι προκαλεί και τι παράγει η γεωργία αλλά και ποιε είναι οι συνέπειες της τοπική οικονομία. Και η επιστήμη και η καινοτομία σίγουρα θα πρέπει να είναι συντροφή μας, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προβληματιστούμε για άλλα θέματα. Γιατί αν δεν ξέρουμε από πριν τι είδου γεωργία θέλουμε και πού θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιστήμη και την καινοτομία, ίσω έχουμε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε, να ζητήσουμε αυτά τα θέματα. Του στόχου μα, τα γεωργικά μοντέλα και αν εξυπηρετούν του οικονομικού περιβαλλοντικού στόχου, τους στόχους της υγείας, ε, της ποιότητας των τροφίμων και από εκεί και πέρα να δούμε αν θέλουμε μια συλλογική προσέγγιση. Και σίγουρα ένα τομέα που χρήζει ε, επένδυσης είναι η δορυφορική τεχνολογία, γιατί εκεί, χάρη στη δορυφορική τεχνολογία, έχουμε τεράστια ακρίβεια χάρη στη δορυφορική τεχνολογία και μπορούμε να δούμε με ακρίβεια τετραγωνικού εκατοστού τι είδους ε, λοιπάσματα χρειαζόμαστε, τι είδους ε, καλλιέργεια χρειαζόμαστε. Και πραγματικά θα πρέπει να έχουμε τα μέσα που μπορούν να μας λένε σε συγκεκριμένο αγροτεμάχιο τι είδους λίπασμα χρειάζεται. Έτσι θα αναχαιτήσουμε αυτή τη φτώχεια του εδάφους. Θα πρέπει όλα αυτά τα νέα μέσα που έχουμε να τα θέσουμε προς, στο, στην εξυπηρέτηση της γεωργίας, της απασχόλησης, της ποιότητας των τροφίμων. Δεν είναι καθόλου απλά τα θέματα. Και η έκθεση αυτή σε τελική ανάλυση αφορά τη συλλογική μας ευθύνη. Σας ευχαριστώ κύριος Σελιμόβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω ολόθερμα τις ε, προσπάθειες του κυρίου Χούιτεμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, διότι η γεωργία πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, προκειμένου να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει βελτίωση λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ευρώ κοινό τη γεωργία και τους γεωργούς. Αν δείτε λίγο τη δημόσια εικόνα του γεωργού στη τηλεόραση, ε, θα δείτε ότι πάντα έρχονται στις Βρυξέλλες ε, και είναι λάστιχα κτλ. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε. Αν πάτε στον κύριο Χούιτεμα και τον ακολουθήσετε ε, και δείτε τι γίνεται στην περιοχή του, ε, θα δείτε πράγματα που δεν φαντάζεστε καν ότι υπάρχουν, διότι δεν τα έχετε δει πουθενά, σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν αντιλαμβάνεστε καν ότι υπάρχει μια τέτοια πραγματικότητα στο γεωργικό τομέα. Και το ευρύ κοινό ε, και το πώς εμπιστεύεται το κλάδο της γεωργίας και τους γεωργούς εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ε, διαμορφώνεται κοινή γνώμη για τη γεωργία. Πρέπει λοιπόν να τη βελτιώσουμε την εικόνα της γεωργίας, πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματική γεωργία και να βελτιώσουμε και την εικόνα του γεωργικού τομέα και των γεωργών. Υποστηρίζω την προσπάθεια, υποστηρίζω σίγουρα ε, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ε, σε κάποιες χώρες υπάρχουν εξαιρετικές πρακτικές, οι οποίες απλώς πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες, χωρίς ε, καν ε, δαπανηρές διαδικασίες και τεχνολογίες. Υπάρχει επίσης και το θέμα των αποβλήτων το οποίο αναφέρθηκε και επίσης να υπάρχει και κάποιο κίνητρο στην νομοθεσία το οποίο θα βελτιώνει και θα προωθεί την αποδοτικότητα του γεωργικού τομέα. Ε, θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ενδεχόμενο το οποίο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη όταν θα γίνει αναθεώρηση της νομοθεσίας, αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ώστε και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του κλάδου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ευρωπαϊκή νότη γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ ε, θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την προώθηση του γεωργικού τομέα και των Ευρωπαίων Γεωργών. Ε, η διατήρηση του βιώσιμου μοντέλου κοινή γεωργικής πολιτικής που βασίζεται στις ε, παραγωγές θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Επίσης, η κατάσταση της αγοράς ε, και λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης ε, σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και όχι στην ποσότητα των προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστούν ε, καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης τα οποία θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους γεωργούς και να διατηρήσουν την ποιότητα της γεωργικής γης και του περιβάλλοντος ως σημαντικός πόρος. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ανευθούμε μέτρα για να ε, δώσουμε ε, αντικίνητρα για τις κάποιες πρακτικές, αθέμητες πρακτικές εμπορίας, μείωση του αριθμού των γεωργών και γυράσκουσα κοινωνία των γεωργών που μειώνει και το γεωργικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να σχεδιάσουμε νέες καινοτόμες χρηματοδοτικές γραμμές για να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση της γεωργίας και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει βιωσιμότητα της γεωργίας, κυρίως αυτές οι οποίες θα εντάξουν και τις νέες γενναίες γεωργών και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε καινοτομίες οι οποίες στόχο έχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω Εκλογήκηση της κατανάλωσης ενέργειας, του ύδατος και άλλων πόρων, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε και την κυκλική οικονομία και να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα και προστασία της βιοπικιλότητας δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε αυτέ τι προκλήσει, διότι μπορεί να εκτεθούμε σε πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε καινοτομία σε όλο το γεωργικό τομέα, από τη βασική γεωργική παραγωγή για τη διατήρηση των υδάτων και των άλλων πόρων, εκλογήκευση τη ε, χρήση ενέργεια ε, και ευφυείς, e e ισορροπημένες και στοχευμένες πολιτικές ε, για την καινοτομία. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με βάση τη βιωσιμότητα και το μέλλον του γεωργικού τομέα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, κύριε Χούιτεμα, για την παρουσίαση που μας κάνατε και θα ήθελα να συμπεριλάβετε όλες αυτές τις συστάσεις στη γνωμοδότησή σας. Σας ευχαριστώ κύριο Α Συγγνώμη κυρία Σένερα. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την πρόταση αυτή και σας ευχαριστώ και για την πρόταση και την παρουσίαση που κάνατε μεν, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινάμε από πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται η παραγωγή για να μπορέσουμε να θρέψουμε όλο τον κόσμο, θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε την Ευρώπη. Και εγώ δεν νομίζω ότι στην Ευρώπη πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή, πρέπει να τη μειώσουμε, διότι υπάρχει κατασπατάληση των τροφίμων, έχουμε μεγάλα πλεονάσματα, ε, αναφερόμαστε σε αναζήτηση αγορών για να απορροφηθούν τα προϊόντα μα. Επομένω, η πρώτη μα σκέψη θα ήταν πώ μπορούμε να εργαστούμε ώστε να μειώσουμε την παραγωγή στην Ευρώπη και να λάβουμε υπόψη και τη ζήτηση ε, για τρόφιμα που διαθέτουμε. Δεύτερον, με βάση και την αλληλεγγύη, διότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνήθως ε, όλοι λέμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά εάν θέλουμε να τους θρέψουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι θα, θα τους στερήσουμε τη δυνατότητα να έχουν την ίδια ε, τη δική τους την γεωργική παραγωγή και να μπορέσουν να αναπτύξουν ε, οικονομική δραστηριότητα και να αναπτυχθούν. Τρίτον, ε, συμφωνώ με πολλά από τα οποία σχολιάστηκαν εδώ και τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της δημόσιας υγείας και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να αναφερόμαστε σε αγροοικολογία, στην διατήρηση των εδαφών και των υδάτων. Ε, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο αυτή τη χρονική στιγμή ε, αναγνωρίζεται σαφέστατα ότι έχουμε φτάσει στο μέγιστο της παραγωγής του πετρελαίου, επομένως θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε μια γεωργία η οποία δεν θα εξαρτάται τόσο από το πετρέλαιο και να δούμε και πώς θα επιβιάσουμε, πώς θα αναζητήσουμε δυνατότητες να μπορέσουμε να ε, χρησιμοποιούμε ε, τροφές ε, για τα ζώα μας τα οποία να μην εξαρτώνται από ε, εισαγωγές γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων και που συνεισφέρουν σε πολλά από προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και σε επίπεδο περιβάλλοντος αλλά και σε επίπεδο παραγωγής. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριλάβετε αυτά τα σχόλια στο εγγραφό σας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη συνεισφορά ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κοινωνία σήμερα και να μην συνεισφέρουμε εμείς στην επιδείνωση των προβλημάτων. Διότι Εάν ε, ληφθούν κάποια μέτρα και χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες οι οποίες απλώς θα δημιουργήσουν περισσότερη ενεργεία και θα συνεχίσουν να παράγονται περισσότερα προϊόντα ε, όταν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε, καλό θα ήταν ε, να το λάβουμε υπόψη και να αλλάξουμε στάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όντως, η δυσκολία έγκυται στο να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ποιότητας ε, της διατροφής, της επικοινομορφίας, της ποσότητας, της, ε, το πώς επηρεάζει την υγεία αλλά και την απασχόληση. Και η σεπήρωση των όσων είπε ο κύριος Ανδρίας θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε και το, τον αγροτικό πληθυσμό, τους γεωργούς, γιατί ε, εξαρτώμαστε από τους γεωργούς και πολύ συχνά είναι πολύ αεροκατοικημένες οι αγροτικές περιοχές, ε, ανάλογα με την ένταση της παραγωγής, ε, της γεωρία και της κτηνοτροφίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια διαφοροποίηση των παραγωγών και των καλλιεργειών, ώστε να έχουμε συμπληρωματικές καλλιέργειες και παραγωγές. Ε, να μην απαγορεύεται να έχουμε ταυτόχρονα και δασοκομεία και κτηνοτροφία για παράδειγμα. Αυτό είναι χρήσιμο και για τον αγρότη αλλά και για τη διαφύλαξη των ισορροπιών μεταξύ των διαφόρων ε, περιφερειών. Ο κύριος Φλάνγκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χόιτεμα, χαίρομαι που είπατε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ε, σε επίπεδο συμβουλίου, αλλά με συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Λίγα πράγματα είναι σημαντικότερα από αυτό, γιατί αφορά τη μελλοντική μας σχέση με τη γη, με το έδαφος. Ε, είναι τεράστια σημασία και αυτό το ξέρουμε όλοι. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να φάμε κάθε μέρα και αν έχουμε ε, ε, τρόφιμα στο τραπέζι μας και φαγητό, αυτό οφείλεται κύριε χάρη στους αγρότες μας. Αναφερθήκατε στα αυτοπαντοποιημένα τρακτέρι, στα drones, είναι πραγματικά συναρπαστικές αυτές οι τεχνολογίες. Ίσως τελικά θα μπορέσει η τεχνολογία να εξασφαλίσει στον άνθρωπο περισσότερο χρόνο ελεύθερο για να μπορεί να εξερευνήσει τον κόσμο και να μην χρειάζεται να εργάζεται 60-70 ώρες την εβδομάδα. Ο φόβος μου είναι όμως, αν δεν ελέγξουμε σωστά τη τεχνολογία, τι μπορεί να κάνει, αν εξήγει του ελέγχου μας, ε, μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση του πλούτου σε ακόμη πιο ολιγομελή ομάδα ανθρώπων. Αυτή είναι η ανησυχία μου και ο προβληματισμό μου, γιατί ενώ πιστεύω ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι θετική, αν τελικά ε, χρησιμοποιηθεί και γίνει η κατάχρησή τη, μπορεί να ωφελήσει μόνο λίγου ε, και αυτό σίγουρα δεν είναι θετικό. Ίσως μπορεί να είναι urban legend αυτό το θέμα της μηχανοποίησης ε, και το πώς έγινε, προχώρησε η βιομηχανία και πόσα, ε, πόσες θέσεις χάθηκαν από τη μηχανοποίηση γιατί ακριβώς ε, δεν είναι τα ρομπότ που θα αγοράζουν αυτοκίνητα ούτε τα drones θα καταναλώνουν, να θα πίνουν γάλα. Δεν είναι λοιπόν χρήσιμο να περιορίσουμε την απασχόληση στη Γεωργία και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτή την ε, επέκταση της χρήσης των ρομπότ. Πού φτάσαμε τώρα στη Γεωργία όποιο, σε όποιον τομέα και αν είναι κανείς δεν μπορεί να βγάλει τα προστοζή χωρίς μία υποστήριξη ή χωρίς επιχορηγήσεις. Ναι, θέλουμε καινοτομία στο μάρκετινγκ, στην εμπορία, καινοτομία στην ε, δημιουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με γεωργικούς συνεταιρισμούς, με ομάδες παραγωγών που θα αξιοποιούν την τεχνολογία αλλά δεν θα εξυπηρετούν τις πολυεθνικές που θα συγχωνεύονται, θα συγκεντρώνονται και θα κάνουν το βίο ακόμη πιο αβίωτο στους γεωργούς. Γιατί όσο και αν καινοτομούν, όσο και αν στην είναι η παραγωγή, αν έχουμε μόνο μία γυναίκα και έναν άντρα που θα ελέγχει 100-200 εκτάρια με τα drones και πάλι δεν θα καταφέρει να, να είναι προσοδοφόρα αν δεν έχουμε καινοτομία. Και εκεί χρειαζόμαστε καινοτομία στην εμπορία, στη θέση τη εμπορία, στην εμπορευματοποίηση γιατί δεν καταφέρουν καν να, βιοποριστούν αυτή τη στιγμή οι γεωργοί, πολλοί γεωργοί. Θέλουμε λοιπόν την τεχνολογία να διευκολύνει τη ζωή των γεωργών. Και σίγουρα το τρακτέρ χωρίς οδηγό δεν θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ζωής στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των αγροτών μας. Γιατί κάτι που μαθαίνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ότι μικρές πόλεις και κομμοπόλεις σαν αυτή τη γενέτειρά μου, εξαφανίζονται από το πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτά όμως είναι τα κοσμήματα και αυτά που ε, δίνουν ε, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο στην, ε, στις χώρες μας, γιατί ωραίες είναι οι μεγάλες πόλεις, αλλά οι μικρές είναι που δίνουν το επιπλέον. Και αυτό φοβάμαι ότι θα γίνει και με την τεχνολογία. Γιατί Φοβάμαι μην απογυμνοθεί η πεθρό μα. Ε, γιατί μιλήσατε κάπως αρνητικά για τι ε, διαμαρτυρίε ε, των αγροτών και των τρακτέρ στους δρόμου. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην πρόοδο, στην γενικότερη πρόοδο τη Γεωργία και όχι να διευκολύνουμε ένα τέρα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτό, να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο ένα τέρα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Σάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική. Είμαι από την Ολλανδία και έχουμε χιλιάδες παραδείγματα καινοτομία στη χώρα μας. Όμως, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οι γεωργοί δεν επιβιώνουν εξαιτίας του κόστους της δουλειάς τους. Χρειάζεται κανείς ε, να βγάζει χρήματα όχι μόνο για να πληρώνει τα έξοδά του, αλλά και για να ζει. Στην Ολλανδία, λοιπόν, γίνεται επεξεργασία στα γαλακτοκομικά, υπάρχουν ε, πολλές ε, τέτοιες δραστηριότητες που, θα, που επιδέχονται νέων λύσεων τις οποίες θα μπορούσε να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να πάμε στο Παρίσι και ε, να συζητήσουμε για την ε, βιώσιμη ενέργεια του 2030, το 2030, ε, θα πρέπει να συζητήσουμε και για τη γεωργία που μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που εργάζονται στον τομέα των βιολογικών προϊόντων ή των εγκαταστάσεων, των γεωργικών εγκαταστάσεων. Πρέπει να συζητήσουμε και για τα λοιπάσματα δεν είναι μόνο η παραγωγή και η ενέργεια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που ε, βοηθούν στην αηφορία. Έχουν να κάνουν με την ηλιακή και ολική ενέργεια, όμως δεν έχουν να κάνουν με την υποβοήθηση άλλων τομέων. Δεν είναι λοιπόν μόνο η καινοτομία. Πρέπει να εξετάσουμε όλους τους τομείς που μπλέκονται και όχι μόνο λίγους εξ αυτών. Ο κύριος Χαϊτόμα έχει και πάλι το λόγο, εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Γι' αυτό ακριβώ ήθελα να γίνει και συζήτηση. Κράτησα σημειώσεις ε, πολλές για τις προκλήσεις που επισημάνατε. Χρειαζόμαστε πόρους που όλο και σπανίζουν στον κόσμο. Θα πρέπει να φροντίσουμε για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και το θέμα της κοινή γνώμης επίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε. Επίσης, βιοπικιλότητα, πολύ σημαντικό θέμα, κλιματικές αλλαγές, απασχόληση ε, ή η ε, ισχύ των πολυεθνικών. Ε, με την καινοτομία θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε νεοφύς επιχειρήσει ή μικρομεσαίες επιχείρησει για να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης και όχι να τις χάνουμε. Και η ακρίβεια ε, είναι σημαντική, η οργάνωση σε επίπεδο αγοράς, η καινοτομία στο θέμα της εμπαρευατοποίησης, οι οργανώσεις των παραγωγών, πολύ σημαντικό θέμα. Και σίγουρα η καινοτομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά και τη γνώση. Και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα πρέπει να βρούμε ε, συνένεση σημείο σύγκληση με του πρασίνου, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τεχνολογία και φύση μπορούν να συμβαδίζουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε πώ ε, ανανεώνεται το έδαφο, πώ η βιοπικιλότητα μπορεί να βελτιώσει τη βελτίωση της ε, να συμβάλλει στη βελτίωση τη βιορική παραγωγή. Μπορούμε να βρούμε σημεία σύγκληση και να αξιοποιήσουμε ταυτόχρονα και τη φύση και τη τεχνολογία. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μακριά και να κάνουμε αλματώδη βήματα πρόοδου. Επίσης, ε, έχουμε δύο πτυχές στο θέμα της ε, κτηνοτροφίας, για παράδειγμα. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καινοτόμα σημεία. Η διαχείριση. Αναφέρθηκα ακροθυγός ε, στην, στην αρχή, στην εισαγωγή, για τα, τις πρακτικές ακριβίας, για τα drones και τη χρήση του στη γεωργία, τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για να αποφύγουμε την υποβάθμιση του εδάφους, πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια κενά με τη γνώση για να μην έχουμε απώλεια θρεπτικών συστατικών και να μην χρειάζεται να, να καταφεύγουμε σε τεχνικά λοιπάσματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την κοπριά. Επίσης να δούμε και τα νέα προϊόντα που θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, που δεν θα χρειάζεται να τα πετάμε για να αποφύγουμε και την κατασπατάληση των τροφίμων και ο κόσμος ζητά πιο υγιεινά τρόφιμα και πιο ποιοτικά τρόφιμα και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Και δεν είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα θρέψουμε τον κόσμο ολόκληρο. Όντω, αλλά μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο για να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο πώ μπορούμε με το πιο αποτελεσματικό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο να παραγάγουμε τα τρόφιμά μα. Και εκεί μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι και μπορούμε και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και όλοι να κερδίσουμε από αυτό. Πολύ σημαντική συζήτηση, πολυεπίπεδη και μπορούμε κοιτώντας το θέμα από πολλά πρίσματα να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο ενθουσιασμός σας ε, και η στράτευσή της ε, θα εξυπηρετήσει αυτή την πολύ σημαντική και εξαιρετική έκθεση. Γιατί η καινοτομία έχει πολλές διαστάσεις, ε, οικονομικές, κοινωνικές και είναι μια λέξη καινοτομία που εμφανίζεται και μερικές φορές ε, ερμηνεύεται πολύ διαφορετικά ανάλογα με τον τομέα. Επίσης ε, θα πρέπει η καινοτομία να είναι φιλική προς τον Γεωργό να βελτιώσει τη ζωή του, να συμβάλλει στην ε, ανάπτυξη της παραγωγής, ε, αλλά στην βελτίωση και της ποιότητας ε, και την ενίσχυση και της παραγωγικότητας. Πολλές προκλήσεις πιστεύω ότι είναι δυνατόν να, τις, να ανταπεξέλθουμε σε αυτές, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απαιτητικοί ότι θα υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους στον ίδιο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. 11 Ιανουαρίου ε, θα συζητηθεί η, η, εκθεση έκθεση. 22-23 ε, Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και 13 Ιανουαρίου η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Πάμε τώρα στο σημείο 8, την απαλλαγή για το 2014, ε, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης ε, είναι ο κύριος Τίμπορ Σάνι. Αρμόδια κατ' ουσίαν για την έκθεση αυτή είναι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, εμείς αποφασίσαμε να στάξουμε γνωμοδότηση για το θέμα της απαλλαγής του 2014 ε, είναι νομίζω προς το συμφέρον μας να εκφέρουμε τις απόψεις μας ε, για το πώς ε, εκτελούνται, εκτελείται ο γεωργικός προϋπολογισμός και το πώς αξιοποιούνται τα γεωργικά κονδύλια. Γιατί ο προϋπολογισμός γεωργίας αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού μαζί με την πολιτική συνοχής. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η σωστή αξιοποίηση των κονδύλιων. Θα πρέπει να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα και θα πρέπει η χρηματοδότηση να γίνεται με διαφανή τρόπο και αποτελεσματικό. Όπως σας είπα, ο εισηγητής, ο συντάκτης γραμματοδότησης μας είναι ο κύριος Τίμπο Σήμερα θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω το λόγο πρώτα στο συντάκτη της γραμματοδότησής μας. Thank you very much, sir. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πάω λίγο πίσω στην προηγούμενη συζήτηση. Ε, σκεμμένα δεν ζήτησα το λόγο προηγουμένως, αλλά στη χώρα μου, στην Ουγγαρία, παλιά είχαμε ένα ωραίο σλόγγαν που έλεγε ότι η ιδιοκτησία θα πρέπει να ανήκει σε αυτούς που την καλλιεργούν. Τώρα, στο σύγχρονο κόσμο, θα πρέπει να λέμε ότι η γη θα πρέπει να ανήκει σε αυτούς που έχουν κατάλληλες γνώσεις, να την καλλιεργήσουν με κατάλληλο τρόπο. Και αυτό σχετίζεται λίγο και με το δικό μου το θέμα, δηλαδή την προετοιμασία για την απαλλαγή του 2014. Ως εισηγητής, συντάκτης μάλλον της γνωμοδότησης, ε, Προσβλέπω στην εξέταση των λεπτομεριών της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για το 2014, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα δημοσιευθεί αύριο. Ελπίζω να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις ε, σε σχέση με τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών και να δούμε πού αλλού θα μπορούσαμε να έχουμε ε, βελτιώσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έκανε σημαντικό έργο το 2014 προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αρχές των κρατών μελών θα μπορούν καλύτερα να προβλέψουν σφάλματα στις γεωργικές δαπάνες, ε, να εφαρμόσουν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου και επίσης ε, ελπίζουμε λοιπόν και εμείς ότι οι προσπάθειες αυτές θα αποτελέσουν ε, καλή βάση για την ε, επταετή περίοδο 2014-2020. Μετά από την ανάλυση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά βεβαίως Πρωτού διαβάσουμε ακόμα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα και θα ήθελα να σταθώ σε τρία εξ αυτών σήμερα. Πρώτον, το 2014 ήταν ιδιαίτερη χρονιά, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ήταν μεταβατική χρονιά. Μεταβατική χρονιά διότι Ε, το θέμα των ε, πράξεων καταξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων διαθετήθηκε μόλις ε, ένα εξάμεινο μετά την έναρξη του 2014, επομένως καθυστερήσαμε στην εφαρμογή. Χρειάζομαι, λοιπόν, χρειαζόμαστε κατανόηση λοιπόν από πλευράς όλων για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεύτερον, Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και τις ε, δραστηριότητες που δεν είναι γεωργικές της κοινή γεωργικής πολιτικής και φυσικά ε, μπορεί να ε, προκύψουν κάποια ζητήματα εδώ. Τρίτον, επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε τις άνισες και υπερβολικές πρακτικές φορολόγησης ε, εν ώψη και της έννοιας των βιώσιμων τροφίμων. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το ελεγκτικό συνέδριο θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην ε, αποδοτικότητα τους επόμενους μήνες και χρόνια, αλλά βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία ασυμμετρία ε, μεταξύ αυτής της προσέγγισης σε, κάποιο, σε ένα χρόνο και ε, την, τον υπολογισμό των δαπανών με βάση αυτά και το πολιετές πρόγραμμα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά και την προσωπική μας επιθυμία ως συνομοθέτες να υπάρχουν ε, προγράμματα τα οποία προσφέρουν κάποια μεσοπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη εξασφάλιση σε όλους όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα διανομής και από τον γεωργό μέχρι τον ε, τελικό καταναλωτή. Και εδώ θα σας μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός της γεωργίας είναι ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά υπάρχουν ε, απλοί λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό. Θέλουμε να έχουμε τρόφιμα καλής ποιότητας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε προσιτές τιμές. Καλή ποιότητα και προσιτές τιμές. Και αφετέρου θα πρέπει επίσης να προβλέψουμε και βιωσιμότητα στο βιωτικό επίπεδο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Θεωρώ ότι μετά από χρόνια και δεκαετίες ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, οι στόχοι αυτοί ακόμα δεν έχουν επιτευχθεί. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο Ζητώ από όλους ε, στην Επιτροπή να κάνουν παρατηρήσεις, ε, προτάσεις ε, για την έκθεση αυτή. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι εξίσου σημαντική σήμερα όπως και στην αρχή για να υπάρχει επιστημιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Και δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε πώς ένας ετήσιος λογιστικός έλεγχος μπορεί να μας δώσει ε, απτά στοιχεία και συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς ε, ε, αποδίδει η γεωργική πολιτική. Και εμείς δεν μπορούμε με αυτά τα μέσα να δούμε πώς λειτουργεί η γεωργική πολιτική. Πέραν αυτού, θα επικεντρωθώ σε τομείς όπου έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές ε, στοιχεία τα οποία έχει εντοπίσει και το συνέδριο, είτε θετικά είτε αρνητικά. Κάποιες πτυχές ε, στις οποίες ε, ακόμα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και επίσης θα επικεντρωθώ σε ευνίδιες αλλαγές το 2014 και το, σε τι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε αυτές τις αλλαγές. Και επίσης υπάρχουν κάποιοι τομείς που με ανησυχούν και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας θα ήθελα να εξετάσουν, όπως για παράδειγμα την, ε, τις διάφορους τομείς που μας απασχόλησαν το 2014 από διαφορετικά οπτικά πρίσματα και όπως έγινε και στην προηγούμενη συζήτηση θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση. Η κοινή γεωργική πολιτική εξακολουθεί να είναι κοινή, εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, ε, σε πεδιάδες, ε, σε ορεινές περιοχές και καλύπτει και φυτίες ε, και ζωοτροφές και τρόφιμα οποιοδήποτε είδους και υπάρχει ο στόχος της συνεχούς υγιούς παραγωγής τροφίμων. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι πιο ουσιαστικά από αυτό να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους κατανοητές και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί πάντα ακόμα και όταν εξετάζουμε τις δαπάνες ε, και τις λεπτομέρειες επί των δαπανών όπως θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες και όταν θα δούμε και τις ε, ε λεπτομέρειες του εγγράφου του ελεγκτικού συνεδρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προσβλέπω στη συζήτηση. Είναι πρώτη ε, συζήτηση όπως είπατε κι εσείς ε, και με τους και συζητητές από τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες θα συζητήσουμε το θέμα της απολογής ε, του 2014 για τη Γεωργία, ώστε να υπάρχει μια άρτια καταρτισμένη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Υπάρχουν ήδη ε, στοιχεία του διαλόγου που έχετε θίξει και τα οποία θα πρέπει να τα ε, αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Καρσέλη έχει πρώτος το λόγο. Ναι, ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ε, όπως επίσης και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, επισημαίνουν ότι τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ε, είναι αποδοτικά από πλευράς κόστου αποτελεσματικότητας. Αν λάβουμε υπόψη τις δαπάνε που γίνονται στον τομέα αυτό, θα δούμε ότι για κάθε ευρώ που δαπανάτε ανακτώνται 40 μέσω των δημοσιονομικών διορθώσεων. Αλλά τα κράτη-μέλη δαπανούν 4 δις για τη διαχείριση και τον έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής που σημαίνει ότι είναι το 7% αυτών που ε, διατέθηκαν το 2014. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρούν ότι οι εθνικές αρχές έχουν περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό και οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2012 και το 2013 διαπιστώνουν ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των διοικητικών ελέγχων και των ε, ε, ελέγχων επιτόπου προκειμένου να βελτιωθεί το η σχέση κόστους ωφελίας και να υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στην κοινή γεωργική πολιτική. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν είναι απαραίτητο να μειωθούν τα σφάλματα και να γίνεται πάντα διάκριση μεταξύ των σοβαρών σφαλμάτων, δηλαδή σφάλματα τα οποία προκύπτουν από ε, ανεπαρκείς ε, πληρωμές ή από υπερβολικές πληρωμές ή απάτες και τα μικρά διοικητικά σφάλματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διακοπή αναστολή πληρωμών σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων και επίσης ότι τα ίσονο σημασία ασφάλματα θα διορθώνονται στην πορεία ώστε να αποφεύγεται ε, να υπάρχουν ε, περιτές ε, διακοπές. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να επισημαίνουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής και η μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Γι' αυτό ακριβώς ε, και η απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, επί της οποίας εργάζεται αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να βελτιώσουμε την εφαρμογή και τη διαχείριση του greening και επίσης για να μειώσουμε ε, το διοικητικό άθος το οποίο επιβαρύνει τους γεωργούς από το 2015 που είναι το έτος ε, ε, που ξεκινά το νέο καθεστώς πληρωμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Εγώ θα επικεντρωθώ στο δικό μου θέμα που αφορά τη χρήση κατάχρηση των πόρων. Την αποτελεσματική διαφανή χρήση των πόρων, την πάταξη της απάτης και τη σχεση κοστος κόστους-οφέλους στους πόρους. Όπως είπατε, ο γεωρικός προϋπολογισμός είναι το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικές φορές αξιολογούνται υπό το πρίσμα της χρήσης ή της κατάχρησης ε, των γεωργικών πόρων. Γι' αυτό και το ζήτημα τη σωστή διαχείριση και εκτέλεση του γεωργικού προπολογισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα ήθελα να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, θα ήθελα να παταχθεί η απάτη, να πιάνουν το, το από περισσότερο τα χρήματα και τα, να βελτιωθούν και τα αποτελέσματα. Τότε δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να δώσω μάχη υπέρ της διαφύλαξης του γεωργικού μας προϋπολογισμού. Είναι θέμα νομοποίησης, ε, είναι θέμα αποδοχής των θεσμικών ε, οργάνων ε, από τον πολίτη, γιατί όσο δεν υπάρχει αποτελεσματική χρήση των πόρων, στο μέτρο που δεν αξιοποιούμε στο έπακρο αυτούς τους πόρους, θα διακυβευτεί και η ίδια η δική μας νομοποίηση, ακόμη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις καταχρήσεις, να αυξήσουμε τη σχέση κόστους-οφέλους και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα του έργου μας. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να υπερασπίσω τους ίδιους πόρους ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριο Φλάνναγκαν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στο σημείο που ο κύριος ε, Σελεμίνοβιτς ανέφερε δύο φορές αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά στην κοινή γεωργική πολιτική. Είναι το να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο που δεν είναι αγρότες ότι αυτά τα χρήματα τελικά πέφτουν και στις, μπαίνουν και στις δικές τους τσέπες. Με αυτό το μήνυμα την διάμεση αναθεώρηση θα καταφέρουμε να κάνουμε και αυτούς που δεν είναι από τη γεωργία να ενδιαφερθούν. Αυτό που προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Εγώ ε, είμαι από μια περιοχή εργατική, ο πατέρας μου ήταν εξυλουργός και η μητέρα μου και όλοι οι άλλοι εκεί ε, ε κριτήκαραν τους γεωργούς ε, και έλεγαν γιατί παίρνουν τόσα χρήματα. Αυτό λοιπόν που στην ουσία πρέπει να τους πούμε είναι ε, ότι κοίτα, εσύ που είσαι ξυλουργός, από πού παίρνει ο ε, αγρότης τα χρήματα για να έρθει να αγοράσει τα δικά σου ε, προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ότι τα χρήματα ε, πέφτουν προς τα κάτω, προς τις κατώτερες τάξεις και δεν ε, πηγαίνουν μόνο στους πλουσίους. Αυτός λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος να, να πουλήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Να μάθει το ευρύ κοινό ότι τα ευρώ δεν πάνε στις τσέπες των γεωργών, ότι ο γεωργός τελικά αυτά τα ευρώ τα ξοδεύει τοπικά μέχρι και το τελευταίο σέντ. Και αυτό είναι όφελος για όλα τα επαγγέλματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό και είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι όλη αυτή η απέχθεια ε, για τους γεωργούς εκτός της γεωργικής κοινότητας είναι περίεργη. Και πρέπει πραγματικά να πουλήσουμε αυτό το μήνυμα ότι τα ευρώ δεν καταλήγουν μόνο στις επιστον των γεωργών και έτσι θα πουλήσουμε και την ΚΑΠ. Ευχαριστώ ο κύριος ο Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας, διότι νομίζω ότι οι πληροφορίες ε, της δικής σας Επιτροπής ε, στην ε, διερευνητική διαδικασία είναι πολύ σημαντικές για να έχουμε μια ισορροπία στην δημοσιονομική διαχείριση αλλά και στις φιλοδοξίες της κοινή αγροτικής πολιτικής. Όπως είπε και ο εισηγητής, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα εκδοθεί αύριο και θα έχει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού την έκθεση αυτή αύριο. Ε, θα ακολουθήσουν εντατικές συζητήσεις εκεί στην Επιτροπή τους με τη δική σας συμβολή φυσικά ε, ε, εμείς επίσης έχουμε μια ακρόαση με τον Επίτροπο ε, στις 14 Ιανουαρίου του 2016. Ως τώρα ε, η Γεωργία αυτά τα θέματα ήταν ένας μοχλός για να έχουμε καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση. Ο περισσότερος έλεγχος ε, για τους γεωργούς ε, σημαίνει και μεγαλύτερες διαδικασίες συμμόρφωσης και αδειοδότησης πριν ε, δοθεί οποιοδήποτε κονδύλι για να μπορούν να χρησιμοποιούνται σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στην έκθεση πεπραγμάτων του 2014 το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος ήταν 2,6% για τον πρώτο πυλώνα και 5,2% για τον δεύτερο πυλώνα. Και θα με εξέπλητε αν τα νούμερα που θα μας δείξουν αύριο από το ελεγκτικό συνέργειο είναι διαφορετικά από αυτά που μόλις σας ανέφερα. Η χρηστή δημοσιονομική πολιτική, όπως είπα, είναι σημαντική, αλλά πρέπει να αντισταθμίζεται και από τα αποτελέσματα και τις πολιτικές φιλοδοξίες μέσα, εντός των πολιτικών. Η έκθεση πεπραγμάτων της Επιτροπής επικεντρώθηκε πολύ σε αυτό που τώρα ονομάζουμε επιδόσεις, απόδοση και ε, εξέτασε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ε, γεωργίας στην Ευρώπη και των μέτρων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βλέπω ότι αυτά ήδη τα ανέφερε και ο συγητής. Ε, δεν αξίζει να δούμε τι συνέβη σε ένα έτος, πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τις πολιετής επιπτώσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής. Μόνο έτσι θα έχουμε ε, μια σωστή και ισορροπημένη κρίση για τις επιδόσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής. Γι' αυτό ε, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις της γεωργικής πολιτικής ε, από την Επιτροπή μαζί με την πρόθεση των αποτελεσμάτων την κυρία Τζεωργίεβα. Είναι πολύ σημαντικό η κοινή αγροτική πολιτική να μην ε, ακολουθεί μία μη ρεαλιστική προσέγγιση και γι' αυτό ακριβώς ανέφερα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την πολυετή προσέγγιση και να μην έχουμε την πιο ε, ε, μηχανιστική και αιτήσια προσέγγιση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Η απλούστευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Όπως ξέρετε, ο Ήτροπος Χόγκαν έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία για την απλούστευση και χρειάζεται την υποστήριξη αυτής της Επιτροπής για να μπορέσει να απλοποιήσει τους κανόνες όπου χρειάζεται χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Πριν λοιπόν καταλήξω να σας δώσω και κάποια στοιχεία περισσότερο ε, αυτά. Αυτή η διαδικασία καλύπτει το 2014, το δημοσιονομικό της 2014 καλύπτεται από αυτή την έκθεση. Ε, όμως αυτό ε, στηρίζεται ε, στις πληρωμές που έγιναν το 2013. Η πρώτη φορά λοιπόν που θα εξεταχθούν και θα κριθούν οι ε, πληρωμές που έγιναν μέσα από την μεταρρυθμισμένη πολιτική θα είναι το 2017. Στα πλαίσια λοιπόν της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής διαχείρισης έγιναν πολλά βήματα. Παρόλο που οι κανόνες και οι οδηγίες ε, γράφονται στις Βρυξέλλες, η εφαρμογή των πολιτικών είναι θέμα των κρατών μελών. Και είναι δύσκολο για την Κομισιόν να διασφαλίσει, να πείσει και να ε, αναγκάσει κάποιες φορές τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την πολιτική, την κοινή γεωργική πολιτική. Όμως πάντοτε η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίζει και γι' αυτό επιμένει ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει ως βασικό στοιχείο της να έχει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και αυτό είναι κομμάτι της απαλλαγής, γι' αυτό ε, ζητώ ε, από την Επιτροπή σας να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και πάλι ο συντάκτης χρηματοδοτησής μας, ο κύριος Σάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ντες. Ε, ήθελα και εγώ να μιλήσω λίγο. Ήθελα να ευχαριστήσω ε, και εγώ τον ε, συντάκτη εκ μέρους της ομάδας μου. Ξέρω ότι ήταν αξιόπιστη η εργασία του και πολύ καλή συνεργασία στο θέμα της γεωργικής πολιτικής. Διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα πάμε ε, σε αυτό το ε, θέμα. Στην, η πιο φτωχή γεωργία είναι στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις στατιστικές υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί γεωργοί στη Γεωργία. Γιατί τα χρήματα που έπεσαν το 50, το 60 και το 70 δόθηκαν για τις υποδομές ε, για, νέες, ε, ε, για νέα εργοστάσια, εταιρείες και λίγο στην εκπαίδευση και Έτσι λοιπόν ε, με αυτές τις επενδύσεις ε, έχουμε 1,6% ανεργία. Ε, αυτή είναι η πιο χαμηλή στην Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταφέρει όλα αυτά. παρόλο που ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση στο παρελθόν, προσπαθούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μας βοηθήσει ώστε σε αυτό ακριβώς το θέμα ε, και στον προϋπολογισμό να προσέξουμε αυτά που χρειάζονται οι συγκεκριμένες περιοχές, αυτές που έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα βρούμε κοινέ ε, λύσεις για αυτό το θέμα. Όσον αφορά στην Επιτροπή, φυσικά εμείς θα υποστηρίξουμε τον Επίτροπο ως Κοινοβούλιο για την μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής. Ξέρουμε ότι είναι πολύπλοκο για διάφορους λόγους, όμως το είπαμε πάρα πολλές φορές ε, και δεν ξέρω αν το είπατε ήδη, ότι αυτή είναι η πρώτη χρονιά της εφαρμογής και πρέπει κάπως, άλλος να, κάπως αλλιώς να το αξιολογήσουμε στον έλεγχο. Ε, να μην έχουμε 100% διόρθωση Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις διοικήσεις στα κράτη-μέλη τον Μάιο και τον Ιούνιο να παίρνουν τις οδηγίες και να πρέπει ήδη το Σεπτέμβριο να εφαρμοστούν. Μπορούν να υπάρξουν προβλήματα και γι' αυτό ε, πρέπει να ε, κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των λάθων που ήρθαν λόγω των λαθών που ήρθαν των οδηγιών και της απάτης γιατί τα λάθη ε, ε, πραγματικά σε αυτό το πρώτο έτος θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με λίγο πιο γενναιόδωρο τρόπο. Σας ευχαριστούμε και τώρα ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ. Από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις που άκουσα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση γιατί θα λάβω υπόψη όλα αυτά τα σχόλια που άκουσα. Και σίγουρα ε, μην ξεχνούμε ότι η αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή δεν είναι η δική μας επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας, αλλά η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, η Επιτροπή που ασχολούνται περισσότερα με το λογιστικό έλεγχο. Πάντως συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι είναι δική μας πολιτική ευθύνη να κοιτάξουμε λίγο και πέρα από τους αριθμούς. Και δεν θα ήθελα να επικεντρωθούμε μόνο ε, στα λογιστικά θέματα και να γίνονται οι βασικές δηλώσεις μόνο από τους αρμόδιους για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Και συμφωνώ κύριε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το περιεχόμενο της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα εντοπίζει υπερβολικά ποσοστά σφάλματος η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Το απέφχομαι, αλλά πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει και γιατί. Με φυσικά βασικό μας στόχο και πρόθεση να διαχωρίσουμε τα λάθη, τα σφάλματα από τις απάτες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ριζική διαφορά. Επίσης, ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μέγκελ, το 2014 ήταν όντως μια ιδιάζουσα χρονιά. Αλλά ήδη βρισκόμαστε στο τέλη του 2015. Και το θέμα αυτό θα διεκπαιρεωθεί γύρω στο Φεβρουάριο του 2016. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα και στους συναδέλφους ε, που θα είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Midterm Review που αναμένεται ως Νούπο. Επίσης, το έργο μας θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ε, αποστολή. Αποστολή μας να διαμορφώσουμε την ε, αντίληψη του κόσμου και για το πώς διάφορες ομάδες της κοινωνίας αντιμετωπίζουν τη γεωργία. Είναι ακόμη παρόν ο κ. Φλάναγκα και θα ήθελα να πω ότι Ε, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν θα παραμείνουν στις τσέπες των γεωργών. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες φημολογίες που κυκλοφορούν και μερικές φορές ακόμη και αποδείξεις ότι αυτά τα χρήματα καταλήγουν όχι στις τσέπες των γεωργών αλλά στις τσέπες της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέξουμε. Και αν θέλετε κύριε αν είστε ευπρόσδεκτος για να συνεργαστούμε και να το ελέγξουμε. Ο κύριος Ελεμόβιτς έφυγε στο μεταξύ, αλλά είπε πολύ σωστά πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να βρούμε το συσχετισμό μεταξύ των δαπανών και της αποτελεσματικότητας. Κατά πόσο δηλαδή πιάνουν τόπο τα χρήματα. Και επίσης ε, συμφωνώ με τον κύριο Βαλκάρσελ θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των σοβαρών σφαλμάτων και των ίσονο σημασία λαθών. Βέβαια υπάρχουν άλλες επιτροπές που ελέγχουν και παρακολουθούν άγρυπνα τα σφάλματα στην εκτέλεση του προπολογισμού. Θα πρέπει πάντως να αλλάξουμε εμείς την εσφαλμένη αντίληψη που έχει ο κόσμος για τη γεωργία. Και αυτή είναι η ευθύνη και το καθήκον μας να διαμορφώσουμε τα μηνύματα για το μέλλον υπό το φως των τεκτενωμένων και το 2014. Και το κλειδί βρίσκεται στη συνεργασία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συμπηλήσουμε όλες αυτές τις ιδέες και σας διαβεβαιώ ότι είμαι πρόθυμος να τις συμπεριλάβω στη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ θερμά για το πολύ φιλικό πνεύμα που δείξατε και ας ανασκουμποθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάνη. Υπάρχει το θέμα φυσικά το πόρων, του τρόπου δαπα, δαπάνης των κονδυλίων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά ε, δεύτερο θέμα είναι η αποτελεσματικότητα τις αξιο... και ο τρόπο που αξιοποιούνται τα κονδύλια. Και φυσικά θα πρέπει να αποφύγουμε και τα λάθη αλλά και τι απάτε και Υπάρχει και το θέμα τη αριστοκρατίας, γιατί μερικέ φορέ τα κονδύλια καταλήγουν εκεί. Τον Νοέμβριο θα υποβληθούν, υποβληθούν οι εξέσεις. 25 Ιανουαρίου θα εγκρίνουμε θα ψηφίσουμε μάλλον για την γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σάνιο ή και θέλει κάτι. Δεν θέλω να είμαι άδικο και ευχαριστώ που το αναφέρατε. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία. το σχόλιο μου ήταν πιο γενικό. γιατί έχουμε και επιχειρηματίες, έχουμε και δικηγόρους, δεν είναι όλοι ολιγάρχες και αριστοκράτες. Απλώς ήθελα να πω όλοι μερικές φορές καταλήγουν σε άλλα χέρια και όχι σε αυτό των γεωργών. Ευχαριστώ λοιπόν 30 Νοεμβρίου για την εξέταση της γνωμοδότησης, 7 Δεκεμβρίου για τις τροπολογίες, κατάθεση τροπολογιών και 25 Ιανουαρίου για την έγκριση της γνωμοδότης. Εξαντλήσαμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη γιατί όπως είπαμε ένα σημείο αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση και το άλλο μεταφέρθηκε στην Πέμπτη. Οπότε ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη στις 12 του μηνός στις 9 το πρωί. Και στις 5.30 σήμερα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι και περιμένω σε λίγο τους συντονιστές. Πεντέμιση ώρα παρακαλώ να είναι παρόντες οι συντονιστές για να περάσουμε στην κυκλισμένο των θερών συνεδριέση. Στους υπόλοιπους σας χαιρετώ. Καλό σας απόγευμα.